Ε, από ευρωπαϊκές πηγές. Πράσινες τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι Σέγγεντη. Τελειώσαμε τη διαδικασία αυτή με τον κύριο Κέλλη του Catch the Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε.